Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νιώθω μεγάλη τιμή που ήσταμε σήμερα ενώπιόν σας ως τμήμα της ομάδος του Jean-Claude Juncker για την Επιτροπή ενώπιον των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των λαών της Ευρώπης, ώστε να ανταλλάξω απόψη μαζί σας, να επιζητήσω την έγκρισή σας για τον διορισμό μου ως Ευρωπαϊκού Επιτρόπου για τα θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για τον εαυτό μου. Ποιος είμαι, ποια είναι η εμπειρία μου και γιατί πιστεύω ότι μπορείτε να μην εμπιστευτείτε. Τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής μου τα πέρασα σε ένα σοβιετικό γκουλάκ, σε ένα γκουλάκ του Στάλιν, στην Βόρεια Σιβηρία, στον Ακτικό Κύκλο. Γεννήθηκα εκεί μέσα σε μια οικογένεια εκτοπισμένων δημοσίων υπαλλήλων από τη Λιθουανία. Όπως ο πατέρας μου, από τα νιάτα μου έχω αγωνιστεί εναντίον της σοβιετικής καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστήριξα πάντα την αλήθεια, την δικαιοσύνη και την ισότητα. Δυο φορές συνελήφθη και ανακρίθηκα από την ΚΑΓΕΜΠΕ. Αγωνίστηκα για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας και είμαι υπερήφανος που είμαι ένας από τις συντάκτες της δήλωσης για την ανεξαρτησία και το σύνταγμα της χώρας μου. Για μένα, ο αγώνας εναντίον του εξτρεμισμού και των ολοκληρωτικών καθεστώτων είναι κάτι το οποίο συνάδει με τη δέσμευση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανθρώπινες αξίες. Υποστηρίζω λοιπόν τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευμάρεια. Και η πολιτική μου φιλοσοφία είναι η σοσιαλδημοκρατία. Δεν έχουμε πρώτη φορά στις Βρυξέλλες. Ήμουν επικεφαλή αντιπροσωπεία τη Λιθουανία στη συνέλευση για το μέλλον τη Ευρώπη υπό τον Ζισκάρ Δεστέν. Ο Τζούλιαν Αμάτο και ο Ζαν Λικ ήταν αυτοί που με δίδαξαν πώς να καταλήγω σε συμβασμούς και συμφωνίες για την Ευρώπη. Γνωρίζω πάρα πολλούς από τους τωρινούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λίγα λόγια στα λιθουανικά. Οι σπουδές μου ήταν στην ιατρική και είμαι καρδιοχειρουργός. Για 23 χρόνια η ζωή μου ήταν να σώζω ζωές ήθελα πάντα να δίνω στους ανθρώπους την ευκαιρία να έχουν μια πιο υγιεινή ζωή. Αυτό είναι το πάθος μου, αυτό είναι η αποστολή μου. Το Μάιο εφέτος εξελέγει αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας. Το άλλο μου πάθος είναι η ιστορία. Σπούδασα την, σπούδασα την ιστορία και έχω ζήσει στο πετσί μου ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας, από τα γκουλάκ μέχρι τον υποψήφιο επίτροπο. Αυτός είναι ο μεγάλος δρόμος για να διατρέξει κανείς σε μια σύντομη ζωή. Είμαι πολιτικός και νιώθω εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια γιατί με εξέλεξαν έξι φορές οι συμπατριώτες μου στην περιοχή του Βίλνιους. Και υπήρξα αναπληρωτής ε, πρόεδρος της Λιθεωνικής Βουλής και Υπουργό Υγεία καθώς και Επικεφαλής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι η υποψηφιότητα μου υποστηρίζεται από το Λουθουανικό Κοινοβούλιο. Τώρα έρχομαι σε ορισμένε από τι προτεραιότητε, οι οποίε θα εστιάσω στα επόμενα πέντε χρόνια. Το να προωθήσουμε την οικονομική ανάκαμψη τη Ευρώπη είναι ένα κέριο στόχο και είμαι πεπισμένο ότι οι πολιτικέ στον τομέα τη υγεία και των τροφίμων, τη ασφάλεια των τροφίμων μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο εδώ. <clears throat> Α ξεκινήσω με το θέμα τη υγεία. Η υγεία είναι ένα βασικό στοιχείο τη κοινωνική οικονομία τη αγορά. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια νέα όθηση για την υγεία στην Ευρώπη γιατί οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι μονάχα δαπάνες. Η έγκαιρη και η παγκόσμια οικουμενική πρόσβαση στην περίθαλψη είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην παραγωγικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε πέραν τη οικονομίστικη άποψη των δαπανών. Πρέπει να δούμε του ανθρώπου και την υγεία του σαν ένα κύριο στοιχείο ενεργητικού για την κοινωνία μα, Γι' αυτό υποστηρίζω τη συνένωση των προσπαθειών των κρατών μελών για να έχουμε περισσότερε επενδύσει στην υγεία και να σώσουμε ζωέ. Μπορούμε από κοινού να κάνουμε περισσότερα, μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα και να βοηθήσουμε του πολίτε μα να ζήσουν πιο υγιεινές ζωέ. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για να του βοηθήσω να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων, ώστε με τον τρόπο αυτό να υπάρξει ισοδύνα, ισοδίκαια πρόσβαση στην ε, περίθαλψη για όλου του πολίτε. Για τον στόχο αυτό θέλω να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα αξιολόγησης που να υποστηρίζει την παγκόσμια, την οικουμενική πρόσβαση στην υγεία, να ενισχύει την πρωτογενή περίθαλψη και να προωθεί την υγεία και την ασφάλεια. Αυτή είναι μερικέ από τους στόχους μου. Οι προτεραιότητες μου λοιπόν για τη δημόσια υγεία είναι πράγματι η προώθηση της ε, υγείας, η πρόληψη και η προστασία. Αλλά αυτό για όλους. Θέλω να ενισχύσω την προληπτική ιατρική. Όσο περισσότερο εστιάζουμε στα υγειονομικά μας συστήματα για την πρόληψη, τόσο λιγότερο θα κοστίσει η θεραπεία σε 10-20 χρόνια. Δεν είμαι εδώ για να σας πω να σταματήσετε το κάπνισμα ή να μην πίνετε. Απλώς θέλω να σας πω πόσο καλύτερη μπορεί να είναι η ζωή χωρίς να καπνίζει κανείς και χωρίς να κάνει κατάχρηση αλκοόλ. η προώθηση μιας υγιεινούς μορφής ζωής είναι μεγάλη σημασία. Αν μπορέσω να αποκομίσω την εμπιστοσύνη σας θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους πολίτες από υγειονομικές κρίσεις ή κρίσεις τροφίμων στο μέλλον. Θα εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη και μπορεί με μεγάλη ταχύτητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση που έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Η επιδημία της έμπολα είναι μια σαφής προειδοποίηση του κινδύνου που μπορεί να προκληθεί από τις λοιμώδεις ασθένειες και τις ανάγκες να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τους πολίτες μας να γεφυρώσουν το χάσμα υγείας στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τις αρχές της ισότητος και της αλληλεγγύης. Υγιή για όλους και όλοι στον σκοπό της επίτευξης καλύτερης υγείας. Τέλο, τέλος θέλω να υπάρξει μια πλήρης εφαρμογή των διαμεθοριακών οδηγιών για την υγειονομική περίθαλψη. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα να υποστηρίξω τα δικαιώματα των ασθενών. Θα παρακολουθήσω επίσης την εφαρμογή της οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα και θα πάρω και τις απαραίτητες ε, μέρημνες για τους εφαρμοστικούς ε, νόμους. Συνεχίζω στα πολωνικά τώρα για την ασφάλεια τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια καλώς ανεπτυγμένη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει όμως να παραμείνουμε επάγρυπνοι και να αντιμετωπίσουμε <clears throat> τις ενδεχόμενες κρίσεις προτεραιότητά μου είναι να εξασφαλίσω ότι οι πολίτες της Ευρώπης θα έχουν τα πιο ασφαλή τρόφιμα στον κόσμο. Χρειαζόμαστε τα ασφαλή τρόφιμα ώστε να εξασφαλίσουμε και την υγεία των πολιτών μας. Τα πρότυπά μας για την ασφάλεια τροφίμων είναι επίσης θετικά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς γιατί μας επιτρέπουν να είμαστε ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές. Θέλω λοιπόν να αξιολογήσω κατά πόσο μπορούμε να απλοποιήσουμε τους κανόνες μας σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων. Ο τομέας αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορεί να συμβάλλει σε μεγαλύτερη ευμάρεια καθώς και σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά του τομέα παραγωγής τροφίμων. Περαιτέρω όμως πρέπει να δούμε και το θέμα των υγιεινών τροφών, γιατί είναι και ένας παράγων από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η υγεία των πολιτών μας. Θα χρησιμοποιήσω κάθε ευκαιρία για να διατηρήσω και να βελτιώσω το σύστημα αυτό, εργαζόμενος με όλους τους εμπλεκομένους. Όλοι έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στο θέμα αυτό, από τους παραγωγούς τροφίμων μέχρι τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Και όλοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Μας έδειξε η πρόσφατη ιστορία ότι μπορεί να υποσκαφθεί η εμπιστοσύνη στα τρόφιμα από τις απάτες και τις κρίσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μειώσουμε το περιθώριο για απάτες και θα υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Μέσα στα πρώτα έξι, μέσα στους πρώτους έξι μήνες της εντολής μου θα ε, περάσω σε μία αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ακολουθώντας τη γραμμή που έχει χαράξει ο Ζαν Κλοντ Ιούγκερ. Επίσης, θα συνεχίσω τις ε, συζητήσεις που έχουν να κάνουν για την πρόταση περαιτέρω καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Επίσης, θα εξετάσω όλες τις προτάσεις που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ιδιαίτερα το πακέτο μέτρων που έχει να κάνει με την υγεία των ζώων, την ε, υγεία των φυτών και τους ε, φυτογειονομικούς ελέγχους που θα πρέπει να ενισχυθούν και συγχρόνως να απλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της καλύτερης ε, νομοθεσίας. Εάν εκλεγώ θα συνεχίσω αυτές τις προσπάθειες με έναν τρόπο ο οποίος είναι διάφανος. Διαφανής. Θεωρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εταίρος μου στα θέματα αυτά. Είμαι έτοιμος να δώσω τις ε, επιλογές που πρέπει να έχουν οι πολίτες μας εδώ και 50 χρόνια αγωνίζομαι για αυτόν τον σκοπό και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Αν έχω την εμπιστοσύνη σας θα εργαστώ μαζί σας που είσαστε οι εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μας και να επιτύχουμε μεγαλύτερη, καλύτερη υγεία. Ξέρουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ας το πράξουμε, ας προχωρήσουμε.